το κόστος των στερεών καυσίμων και του φυσικού αερίου θα είναι τριπλάσιο. Και μετά οι καταναλωτές λένε πώς επιτρέπεται να ε, καταστρέφεται η αλληλεία και ο τουρισμός και τώρα κάνατε αυτά τα ελληνικά πάρκα και τριπλασιάστηκε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Για ε, και εκ των υστέρων χρειαζόμαστε ε, πολύ περισσότερες προσώτες από ό,τι στις κλασικές μορφές ενέργειας. Συγγνώμη που είμαι τόσο επικριτικός, αλλά έχουμε εδώ να κάνουμε με ένα πραγματικό σκάνδαλο. Και εμείς ε, εδώ στην Ευρώπη τι κάναμε. Ζητήσαμε με οποιοδήποτε τίμημα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς να σκεφτούμε ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις. Απ' την άλλη τώρα, η άλλη πλευρά του νομίσματος. Εξετάσατε τις εργασίες που μελετήσατε που έγιναν για την κατασκευή αυτών των εγκαταστάσεων οψών για την δημιουργία Can encourage των πεδίων αναπαραγωγής ε, διότι σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις που είχαμε ε, υπεραλίευση μπορούμε να έχουμε τώρα τέτοιου είδους παιδί αναπαραγωγής Και ίσως αυτό θα ήταν μια ευκαιρία την οποία δεν θα πρέπει να χάσουμε εάν προχωρήσουν στην κατασκευή τέτοιων εγκαταστάσεων offshore. Από τη δική μου άποψη αλλά είναι η προσωπική μου, δεν θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν συμφωνώ. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ ως πρόεδρος έκανα τις πρώτες ερωτήσεις, υποφελήθηκα και ζητούν τώρα και άλλοι συνάδελφοι το λόγο. Κυρία Λέβιν. And uh, thank you very much. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Ε, είναι πολύ θετικό που μας λέτε ότι προχωρούν τα σχέδια για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε λίγα περισσότερα σε ό,τι αφορά τις ε, αξιολογήσεις αντικτύπου αν υπάρχουν, λογικά εσείς θα γνωρίζετε ποιος θα μπορούσε να είναι ο αντίκτυπος αυτών των αιωλικών πάρκων ε, στην ε, αλληλεία, στα ηχθιαποθέματα γενικά, στη βιοπικιλότητα και επίσης ε, στα πτηνά. Γιατί και αυτό θα ήταν ενδιαφέρον. Και να σχολιάσω κάτι στα όσα είπε ο Πρόεδρος για το κόστος. Βεβαίως, το αρχικό κόστος θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο ε, σε ό,τι αφορά τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε σχέση με τα κλασικά καύσιμα. Αλλά βεβαίω υπάρχουν και πολλές επιχορηγήσεις και θα υπάρξουν και οι επόμενες ε, γενιές. Επομένω, δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε με τέτοιο τρόπο. Πρέπει να έχουμε μια οπτική που να αφορά περισσότερο το μέλλον. Αυτά τα ερωτήματα είχα να θέσω στον ομιλητή. Ευχαριστώ. Vorsitzender. Äh, äh, Σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση που ακούσαμε. Άκουσα από κάποιο συνάδελφο ότι έχουμε επιστρέψει στη δεκαετία του 80. Γιατί υπάρχει μια περιοχή με ολικά πάρκα και ε, ακούμε όλα τα επιχειρήματα ε, και στο τέλος είμαστε όλοι πάρα πολύ περήφανοι από τις νέες εγκαταστάσεις και 30% της ενέργειας που χρησιμοποιούμε ε, δημιουργείται, παράγεται από αυτές τις αιωλικές εγκαταστάσεις. Ε, είδαμε όμως τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιαπωνία και βλέπετε ότι η κατάσταση είναι πολύ περίεργη. Μήπως βρισκόμαστε στην σωστή ε, χρονική στιγμή υπάρχει σχεδιασμός και στην ε, Βαλτική θάλασσα και στην Βόρεια θάλασσα, αλλά και οπουδήποτε αλλού υπάρχει δυνατότητα. Και αν δεν έχουμε το σωστό σχεδιασμό θα καταλήξουμε σε ένα χάος. Και όπως υπογράμμισε και ο κύριος Στίβενσον, δυστυχώς εγώ σήμερα ε, τρέχω από συνεδρία σε συνεδρίαση και δεν άκουσα την εισαγωγή της συνεδρίασής σας. Ίσως λοιπόν έχω χάσει κάποια βασικά πράγματα. Ε, αλλά θα ήθελα να πω σε ό,τι αφορά αυτόν τον ε, χωροταξικό θαλάσσιο σχεδιασμό τι έχει γίνει. Ε, εγώ έχω, συζήτησα πρόσφατα με κάποιους αλληλείς και ε, μου είπαν ότι φοβούνται, ανησυχούν, φοβούνται ότι τα δικά τους τα συμφέροντα δεν θα ληφθούν υπόψη ε, δεν πρέπει λοιπόν να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Πρέπει να σιγουρευτούμε ότι θα συνεργαστούμε με τα ε, ενδιαφερόμενα μέρη, με όλους τους εμπλεκόμενους. Και πρέπει να δούμε ποιος επακριβώς είναι ο στόχος, ε, ο αντίκτυπος αυτών των ολικών πάρκων.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 δούμε τι γίνεται στο τομέα της με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις επιπτώσεις την ηλεκτρική ενέργεια, βλέπουμε ότι η τάση είναι να στραφούμε από τις εθνικές αρμοδιότητες προς τις κοινοτικές. Όχι διότι θέλουμε να εμπιστευτούμε συμπληρωματικές αρμοδιότητες στην Ευρώπη, αλλά για λόγους ασφαλείας της προμήθειας ή για λόγους που αφορούν τον ανταγωνισμό και την πρόοδο στις αγορές. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν χρειαζόμαστε διασυνοριακά να κάνουμε ε, ανταλλαγές για την ηλεκτρική ενέργεια πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα. Εξάλλου υπάρχει και η σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει ότι για λόγους ασφάλειας του ανεφοδιασμού και για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας θα πρέπει να υπάρχει διασυνοριακός ποσοστό ανταλλαγών ε, σε επίπεδο 10%. Και το Ηνωμένο Βασίλειο στο μέλλον θα αποτελέσει συμβαλόμενο μέρος αυτής της ευρωπαϊκής ε, ε, ενεργειακής αγοράς μέσω καλωδίων. Διότι αν δεν έχουμε ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό δίκτυο δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε ε, δυσκολίες όπως αυτές που αντιμετωπίσαμε πέρσι το χειμώνα. Εάν το δυναμικό που μπορούμε να αναπτύξουμε είναι 350.000 γιγαβάτ στην Βόρειο Θάλασσα και δεν το εκμεταλλευτούμε, αυτή τη δυνατότητα που μας προσφέρεται. Όταν δεν φυσάει ο άνεμος, θα πρέπει να μπορούμε να προσφύγουμε σε άλλες ε, μορφές ενέργειας για να μπορέσουμε να έχουμε αποθέματα που θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε μετά 24 ώρες, 24 ώρες σε περίπτωση ανάγκης. Θα πρέπει λοιπόν όλο αυτό το σύστημα δικτύο να είναι ασφαλές 2020 και 2030 χρειαζόμαστε 42.000 μέτρα ε, γραμμές υψηλής τάσης συμπληρωματικές στην Ευρώπη για να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα διότι θα πρέπει να προβλεφθούν ε, αυτές οι γραμμές υψηλή τάσεως σε μέρη που δεν θέλουμε να τα έχουμε δυστυχώς. Είναι όμως ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικές οι επενδύσεις σε οι πολύ καλά δίκτυα και σε δίκτυα επιδόσεων. Τώρα όσον αφορά τις κοινωτικές αρμοδιότητες. Εγώ ανέφερα το άρθρο 104 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Τα κράτη-μέλη όμως θα πρέπει να οργανωθούν για την δική τους παραγωγή ενέργειας. Όσον αφορά το ενεργειακό μείγμα, την επιλογή δηλαδή που θα κάνουν, κάθε χώρα μπορεί να επιλέξει πώς θα παράγει την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται. Απ' την άλλη μεριά όμως, οι διάφορες χώρες δεσμεύονται το στόχο του 20%. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιό Γνωρίζουν ότι υπάρχουν τα εθνικά προγράμματα δράση για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το στόχο αυτό τα κράτη-μέλη. Στα πλαίσια αυτών των προβλημάτων προβλέπεται η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ των οποίων σε πολύ καλή θέση βρίσκεται η ολική ενέργεια. Τώρα, θα πρέπει να εγκαθίσετε τα αιωλικά πάρκα κοντά στις ακτές ή ε, πιο μακριά. Αυτό είναι θέμα απόφασης κάθε κράτους. Διότι αν πρέπει να αποφασίσει και για αυτά τα θέματα και να νομοθετήσει η Ευρώπη, δύσκολα οι αποφάσεις της θα γίνουν αποδεκτές. Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, επιμένω στο γεγονό ότι υπήρξε απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης πέρσι να χορηγηθούν τρεις σημαντικές άδειε στη Βόρεια Θάλασσα. Και οι άδειε αυτές αντικατοπτρίζουν τη λύση της απομάκρυνσης από τις άδειε. στην Σκοτία, στην Αγγλία και στην, ε, ε στην Ουαλία. Όσον αφορά την αξιολόγηση των επιπτώσεων, που τέθηκε προηγουμένως από πολλούς βουλευτές, να ξενοποιούμε και από την κυρία Ρόντουστ, όταν έχουμε να κάνουμε με κατασκευή αιωλικών πάρκων, εφαρμόζουμε τις διάφορες σχετικές οδηγίες για τα οικοσυστήματα, την προστασία της χλωρίδας, της πανίδας, της, ε, των ε, αδειών για την κατασκευή των νεολικών πάρκων και για την εγκατάσταση των καλωδίων πάντα θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να γίνουν σεβαστές ε, κάποιοι, σεβαστοί κάποιοι κανόνες για να προστατεύεται γενικότερα το περιβάλλον και η χλωρίδα και η πανίδα. Και βεβαίως πάντα θα πρέπει να γίνονται σχετικές μελέτες επιπτώσεων και ο αντίκτυπος και στους αλληλευτικούς πόρους. Προβλέπονται λοιπόν διαδικασίες για να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγις τι ακριβώς ε, γίνεται. Και βεβαίως ισχύουν οι νόμοι και οι κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος ακόμη και αν κανείς απομακρύνεται από τις ακτές. κυρία Ρόντοστ επίσης αναφέρθηκε στο θέμα της ε, ενέργειας πέραν των συνόρων και είπε ότι η περιοχή της είναι περήφανη διότι 30% της ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της παράγεται από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Σωστό αυτό, αλλά αυτό το οποίο είναι πιο σημαντικό είναι να δούμε τι αποτελέσματα θα μπορέσουμε να έχουμε σε επίπεδο Ευρώπη. Και ελπίζω ότι χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας θα ξεπεράσουμε αυτά τα ποσοστά και θα έχουμε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγαλύτερα ποσοστά από ανανεώσιμες. Επίσης ξέρουμε ότι εκτός από την ε, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να δούμε πώς θα λύσουμε και το πρόβλημα της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θα πρέπει τώρα να γίνει η διαφοροποίηση μεταξύ των επενδύσεων που γίνεται στα αεολικά πάρκα όπου χορηγούνται σημαντικά βοηθήματα και δίνονται επιδοτήσεις βάσει ενός προγράμματος που τέθηκε σε εφαρμογή από πέρσι, αλλά υπάρχουν και τα δίκτυα και σίγουρα ο κύριος Έτιγκερ θα κάνει και προτάσεις για αυτό το τελευταίο θέμα. Δεδομένου ότι θα πρέπει η προσέγγιση μας να βασίζεται και στα κεφάλαια που μπορούν να διατεθούν. Διότι υπάρχουν και θέματα τα οποία αφορούν και τις ε, επιδοτήσεις αλλά και, τους, ε, και τα δημόσια κονδυλώσεις αναφορά την ε, Σκοτία κύριε Πρόεδρε. Ο συντονιστής Εγώ δεν θέλω να εκφράσω τη δική μου άποψη για θέματα που δεν είναι της δικής μου αρμοδιότητας. Εγώ είμαι σε διαρκή επαφή με τον ε, υπουργό σας και οι συζητήσεις στο επίπεδο της κυβέρνησης της Σκοτίας είναι πολύ ενδιαφέρουσες για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς στην περίπτωση της ε, δικής σας ε, εμπειρίας να γίνει κάτι το οποίο θα αποτελέσει πρότυπο κατά κάποιο τρόπο. Και υπάρχει και η δυνατότητα χρησιμοποίησης του παλιροϊκού κύματος διότι και εκεί υπάρχουν δυνατότητες που μπορεί κανείς να εκμετατευλευτεί και όχι μόνο για να καλύψει τις ανάγκες της σκοτίας, αλλά και περαιτέρω. Εγώ τουλάχιστον στο Εδιμβούργο που επισκέφθηκα 4-5 φορές είδα να υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν κάποιες εντάσεις όσον αφορά τη θέση του Λονδίνου, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ δεν είμαι πολιτικός, εγώ είμαι συντονιστής θα έπρεπε να πω ότι αυτό που προτιμώ στη Σκωτία είναι το ουίσκι και όχι οι ολικές φάρμες. Μια σύντομη παρατήρηση. Κύριε Αμπράμοβιτς, θυμήσατε το τι σημαίνει το Σλέβιν Χόλσταϊν. Δεν θέλω να προωθήσω τον περιφερειακό χαρακτήρα, αλλά να πειράξω λίγο τον κύριο Στίβενσον, γιατί αυτά που είπε μου θυμίζουν λίγο αυτά που λέγαμε στους συντηρητικούς συναδέλφους μας ε, στο 1980, οι οποίοι είναι πολύ ικανοποιημένοι από αυτά που μεσολάβησαν στο Σλέβι Χολστάιν. Η αναφορά στο περιβάλλον είναι κάτι το αυτονόητο πλέον βέβαια υπάρχουν ε, συγκεκριμένοι κανόνες και νόμοι που είναι σε ισχύ. Αυτό το οποίο είναι λιγότερο προφανές όμως και σε αυτό καταλήγω ακούγοντας αυτά τα οποία ισχυρίζει το Στίβενσον και δεν είναι μόνος άλλωστε, είναι το θέμα της ε, συμμετοχής των ενδιαφερομένων, των εμπλεκομένων, οι οποίοι θα πρέπει, των οποίων η φωνή θα πρέπει να ακούγεται και δεν συμβαίνει αυτό πάντα. Ίσως να έχουμε συζητήσει με ορισμένους από τους εμπλεκομένους, αλλά αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν έχουν ερωτηθεί, τότε αυτοί είναι φυσιολογικό να καταφέρονται εναντίον του προγράμματος αυτό. Πρέπει να τους πείσετε για να είναι ε, ε, μαζί σας. Θα απαντήσω ευχαρίστως στην παρατήρησή σας. θα πρέπει να δούμε το πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να πείσουμε. Δηλαδή εδώ είναι σημαντικός ο ρόλος των περιφερειακών αλλά και των τοπικών ε, αρχών. Είναι αλήθεια ότι η αλληλεία είναι ένας τομέας πολύ σημαντικός στη Βόρεια Θάλασσα. Δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Και σχετικά με αυτά που είπατε για το ουίσκι κύριε Στίβενσον δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας. Σας ευχαριστώ γι' αυτό κύριε οι κάτοικοι της δικής μου εκλογικής περιφέρειας θεωρούν ότι αγνοήθηκαν στα πλαίσια αυτά της συζήτησης, πάντως είχε ενδιαφέρον και ήταν πολύ καλή η παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλώς, λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε στο επόμενο θέμα. Είναι η συνάντηση των ε, συντονιστών. Η επόμενη συνάντησή μας, η επόμενη συνεδρίασή μας της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής είναι 24η Μαρτίου από τις 3 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα και 24 από τις 9.30 ε, το πρωί μέχρι τις 12.30. Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε, ολοκληρώνεται η συνεδρίασή μας σήμερα και νομίζω ότι οι περισσότεροι από τους συντονιστές είναι ήδη εδώ. Θυμίζω ότι η συνεδρίαση των συντονιστών γίνεται και κλεισμένων των θυρών. Γι' αυτό παρακαλώ όλους τους άλλους παρισταμένους και ε, να αποχωρήσουν.